Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε περάσει 4 ώρε. Να συνεχίσουμε με το σημείο 5. Έχω την ικανοποίηση να καλωσορίσω τον κύριο Γέρζη Παμιανόσκη, τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, για να μα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του Ταμείου για το 2018. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο τη Δημοκρατία λειτουργεί από το 2013 και ήταν πολύ ενέργο αυτά τα πέντε έτη λειτουργία υποστηρίζονται όσου χρειάζονται υποστήριξη σε πάνω από 700 πρωτοβουλίε, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ αξίας και έχει κερδίσει τη φήμη ε, μιας οργάνωσης ε, που επηρεάζει τα πράγματα στις δημοκρατίες. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο που παρουσίασε την ετήσια έκθεση και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που με δίνετε. Για όσους ε, δεν έχετε αντίγραφο PDF ε, υπάρχει και ένα ε, αντίτυπο τυπωμένο στην αίθουσα. Πρόκειται για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία και τις σχετικές δραστηριότητες για το 2018. Καθώς κάνουμε αυτή την παρουσίαση σε τήσια βάση ήδη εδώ και πολλά χρόνια, είναι ιδιαίτερα προνομιούχος η κατάσταση που χαίρει η οργανωσή μου. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα εννέα μέλη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο του Ταμείου συμμετέχουν στη στρατηγική καθοδήγηση του Ταμείου. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω το γεγονός ότι το Ταμείο συχνά αναφέρεται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παίρνει το χάρη σε ένα που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ένα μελλοντικό δρόμο για την περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοαφρική, όπου ζήτησαν τα κράτη-μέλη να συνεχίσει η υποστήριξη στο έργο μα. Η γραμματεία του Ταμείου, που αποτελείται από μια πολυεθνική ομάδα έχει δεσμευτεί για να υλοποιήσει την αποστολή μας και να υποστηρίξει τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Επιτρέψτε μου να φέρω στην προσοχή σας τέσσερα κύρια μήνυματα της έκθεσης. Καταρχήν, πέρσι, το 2018, ήταν ε, το πέμπτο έτος λειτουργίας ε, της δράσης μας και είχαμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γιορτάσουμε και την πενταετή μας επέτειος η πέμπτη επέτειος ε, γιορτάστηκε εδώ και έδωσε κάποια εμπνευστική ευκαιρία για να εξετάσουμε αναδρομικά τη λειτουργία του Ταμείου. Βάσει πολλών σχολείων που λάβαμε, το Ταμείο έχει αναγνωριστεί και έχει γίνει ένας αναγνωρισμένος μηχανισμός για τη δημοκρατία και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Και όπως είπα, ε, αναφέρθηκα στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, όμως ε, και η Κομισιόν και άλλα θεσμικά όργανα ε, έχουν επιτυχώς εφαρμόσει το μοντέλο τους ε, στο κεφάλαιο αναδρόμησης της, ε, της θα βρείτε ε, κάποια αριθμητικά στοιχεία πάνω από 5.000 αιτήματα για υποστήριξη έχουμε λάβει και 722 επιχορηγήσεις συνολικά 50 εκατομμυρίων ευρώ έχουν χορηγηθεί το ταμείο ε, βασίζεται σε καθημερινές δραστηριότητες. Ε, θα σας παρουσιάσω ένα παράδειγμα. Το περασμένο μήνα επισκέφθηκα τα ψήπεδα του Γκολάν, ένα δικαιούχο. Είχαμε ένα ε, ξεκάθαρο παράδειγμα υποστήριξης, καθώς δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει οικονομική στήριξη λόγω των κατεχόμενων καθεστώτος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στη Ρωσία, όπου πολλοί δωρητές για πολλούς λόγους αποφύγουν από την ε, άμαση υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων και είναι προφανεί οι ανάγκε και σχετίζονται με, το με τη μελλοντική ασφάλεια τη Υπήρου μα. Από την έννοια αυτή, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που διαβάζουμε στην πρόσφατη έκθεση της Άννα Φωτίγκα για την ε, στρατηγική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αναφέρεται το Ταμείο και το έργο του ως ένα καλό παράδειγμα για τη δημιουργία ενός πιο πλουραλιστικού περιβάλλοντος ε, στα ε, ρωσόφωνα μέσα. Θα ήθελα να τονίσω το έργο μας για το 2018. Η έναρξη ε, δημοκρατικής ε, ενέργεια στην Αρμενία υποτέλεσε μια έμπνευση για μας. Τα κινήματα των πολιτών ε, και τα κινήματα της αντιπολίτευσης μπόρεσαν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των ε, Αρμενίων συναντήσαμε νέους που έπαιξαν ε, έναν εξέχοντα ρόλο στις διαδηλώσεις που ήταν ειρηνικές και με καλή διάθεση. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία ε, της κοινωνίας των πολιτών στην Αρμενία γιατί ε, μπόρεσε να διαχειριστεί αυτές τις μαζικές ε, διαμαρτυρίες με έναν ειρηνικό τρόπο, αν και υπήρξαν απόπειρες ε, να υπάρξουν βιοπραγίες. Η επέκταση της δράσης μας στην Τουρκία και στα Δυτικά Βαλκάνια, τα βρίσκεται αυτά στις σελίδες 30 και 50-51, ήταν επίσης σημαντικό βήμα για μας. Και πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για νέες δραστηριότητε του Ταμείου, όπω βασίστηκε από το Συμβούλιο μας μόνο πριν 1,5 έτος. Έτσι λοιπόν, ε, μόνο ένα χρόνο λειτουργούμε και το 2018 ήταν το πρώτο έτος δράσεων μας εκεί στην Τουρκία. Βλέπουμε ε, τον αντίκτυπο του έργου του Ταμείου και το περιβάλλον, ε, ενώ το περιβάλλον γινόταν πιο κατασταλτικό και αποσύρονται άλλοι δωρητές. Εδώ η υποστήριξη του Ταμείου ήταν σημαντική για να επιβιώσουν εξάρτητα μέσα ενημέρωση, καθώ και για την δημιουργία νέων οργανώσεων υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστηρίζουν του δημοσιογράφου, όπω ε, η Ένωση για την Ελευθερία ε, του Λόγου. Στην Αίγυπτο συνεχίσαμε το σημαντικό έργο μα να υποστηρίξουμε οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα δίκτυά του. Πολλέ από αυτέ υπέστησαν ε, άμεση δίωξη και καταστολή από τι αρχέ. Και θέλω να καλωσορίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωβουλευτέ επιτυχούν ευτυχώς ε, έχουν παρέμβει για να υποστηρίξουν τους εταίρους μας ε, όταν χρειαζόταν στην Τινησία. Οι εταίροι του Ταμείου εργάστηκαν ε, για να βοηθήσουν το νεοελεκθέν Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις τοπικές εκλογές και το Συμβούλιο θέλει να απαντήσει στα αιτήματα των ε, πολιτών. Είναι ζωτικό να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε την πίστη στη δημοκρατία. Στην ε, Μολδαβία το Ταμείο υποστήριξε ε, ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι όταν μπλοκαρίστηκε η αδειά του και κανένας άλλος δωρητής δεν ήταν έτοιμος να λάβει το κίνδυνο. Επίσης το Ταμείο έπαιξε ζωτικό ρόλο στον να υποστηρίξει το Pro TV και το Journal TV όταν υπέφεραν από Εχθρική νομοθεσία και κατασταλτικά μέτρα. Αυτέ είναι τρει ανεξάρτητε τηλεοράσει ε, εθνικού βεληνικού στη Μολδαβία. Αν ε, είχαν υποστεί καταστολή, τότε θα υπήρξαν σοβαρέ συνέπειε. Ό,τι αφορά την Ουκρανία, ξέρω ότι πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ στην Ουκρανία τουλάχιστον και μετά τις χθεσινές εκλογές. Ε, η μεγάλη ανησυχία μας ε, για όλο το έτος του 2018 ήταν ότι αυξάνονταν ε, οι φυσικές επιθέσεις, σωματικές επιθέσεις και πυροβολισμοί και μαχαιρώματα κατά ακτιβιστών που δρούν κατά της διαφθοράς σε πάρα πολλές πόλεις, στην Οδύσσο και στην ε, Μαριάνοπολ. Έχουμε πάνω από 50 τέτοιε περιπτώσεις. Είναι ενισχυτάση αυτή και δείχνει την αδυναμία του κράτους στην Ουκρανία και την ανικανότητά του να προστατεύσει του ξεδιστέ και να διώξει τους δράστες. Ε, από την άλλη πλευρά όμω, φαίνεται η αποτελεσματικότητα τη ε, ακτιβιστική δράσης των πολιτών και είναι τόσο γνωστή στους κακούς που διευθύνουν ε, τις ε, δομές που εκτίθενται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προβαίνουν σε σωματικές επιθέσεις. Στην έκθεση αποφασίσαμε να φερώσουμε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για το ρόλο των γυναικών και των νέων σε προγράμματα υποστήριξης της δημοκρατίας. Συνεχώς αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντική εταίρη στην επίτευξη ισότητα για τι γυναίκε Στη σελίδα 48 παρουσιάζουμε δύο πρωτοβουλίε ε, στο Μαρόκο και στη Συρία. Επίσης, να τονίσω το έργο μας με ακτιβίστριες στην Μολδαβία. Μετά τις πρόσφατες εκλογές στη Μολδαβία, κοινοβουλευτικέ εκλογές, Είμαστε πολύ περήφανοι που βλέπουμε έξι νέα μέλη γυναίκες του Κοινοβουλίου. Όλες ε, ήταν ακτιβίστριες σε πρωτοβουλίες που υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο. Όπως βλέπουμε και σε πολλέ άλλε χώρε ε, παραδοσιακή πολιτική συζήτηση ε, συχνά είναι καλοπιστική. Όμως ε, συχνά υπάρχουν πρωτοβουλίες ε, των πολιτών. Και επίσης είμαστε περήφανοι που πολλά χρόνια πειραμάτων και δοκιμών κατέληξαν τώρα στην έννοια της, ε, του νέου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης ε, που εισάγει το Ταμείο. Αυτό είναι σημαντικό τμήμα της μεθοδολογίας μας, δηλαδή παρέχοντας επιχορηγήσεις και παρακολουθώντας πώς αναπτύσσουν οι εταίρες μας ιδέες, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση είναι ε, ε, κομμάτι που ανήκει στο ΙΔΙ e και δείχνει όχι μόνο τον αντίκτυπο του έργου μας, αλλά μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς την προσέγγιση μας βάσει των διδαγμάτων. Σελίδα 54 και 55. Εκεί βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό και ανυπομονούμε με τα κράτη-μέλη να συζητήσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας και φυσικά το πράττουμε αυτό όταν θα έχουμε και την ευκαιρία και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις αντίστοιχες επιτροπές αν προσκληθούμε. Ένα πρόσθετο σχόλιο στο στάδιο αυτό. Όπως αναφέρθηκε και πριν, το Ταμείο έχει γκρίνει περίπου 750 επιχορηγήσεις. Όμως υπάρχουν και πολλές απορρίψεις ε, από τις 5.000 αιτήσει. Είναι αναπόφευκτη η κατάσταση αυτή. Πολλοί ε, ετούντες που απορρίφθηκαν μας είπαν ότι έχουν φίλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είδαμε αύξηση τέτοιων περιπτώσεων αφού ξεκινήσαμε το έργο μας στα Δυτικά Βαλκάνια, παραδείγματο χάρη. Ελπίζουμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα κατανοήσουν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την εντολή μας και να συνεχίσουμε ε, να ε, συμπληρώνουμε το έργο άλλων δωρητών και δεν μπορούμε να καλύψουμε κάθε μία αίτηση παρόλο που θα το θέλαμε. Και τέλος, καταληκτικά θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια που επίσης βασίζονται στο έργο που διήρκεσε πάνω από ένα έτος να αναφέρω κάποιες σκέψεις για την υποστήριξη της δημοκρατίας στην Ευρώπη, ιδίω όταν έχουμε νέα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Δημοκρατία υπό εκπόνηση. Αυτά βασίζονται στην εμπειρία μας. Βλέπουμε και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε δύο τέτοιες εμπειρίες και συμβουλές. Πιο συγκεκριμένα, συστήνουμε να υπάρξει μια νέα σειρά κανόνων που θα επιτρέψουν ε, ταχύτερα και ίσως αυτόματα την επακατανομή των κονδυλίων σε περίπτωση που μια σημαντική χώρα εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, έχει συνάψει συμφωνία με τη Σύμβαση ε, διότι ότι υπάρξει ε, σημαντική επαναχώρηση στα δημοκρατικά πρότυπα. Είδαμε παραδείγματα Αζερβαϊτζάν, Αίγυπτος, Τουρκία τα τελευταία χρόνια που κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών επιδεινωνόταν μέσα σε εβδομάδες παρά σε μήνες. Στην χειρότερη περίπτωση ελπίζουμε να μην γίνει, αλλά μπορεί να το δούμε και στη Μολδαβία. Η ιδέα είναι ότι τα εφιστάμενα κονδύλια αυτόματα ε, που δεν έχουν δαπανηθεί αυτόματα να δοθούν ε, στα ανεξάρτητα μέσα της κοινωνίας των πολιτών και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, κατά κάποιο τρόπο το Ταμείο συμμετέχει σε προσπάθειες να υλοποιηθεί με τέτοια προσέγγιση, παραδείγματος χάρη με το διαχειρισμό των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Τουρκία, Αίγυπτο, Αζερμπαϊζάν. Σήμερα όμως ε, είναι σε πειραματικό στάδιο αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί έναν μηχανισμό. Αυτό αποτελεί μια ποικιλομορφία της ρεσιμότητας λιγότερα για λιγότερα. Και θέλουμε να το μεταμορφώσουμε σε more for more, σε περισσότερα για περισσότερα για την κοινωνία των πολιτών. Κάτι ακόμα που θέλουμε να προσθέσουμε, να κατανοήσουμε αυτό που ονομάζουμε υβριδικές απειλές συχνά. Οι υβριδικές απειλές αποτελούν ένα σύνολο θεμάτων, παραπληροφόρηση, ψευδοειδήσεις, ψευδής κοινωνία των πολιτών, διάφορες χειραγωγήσεις. Και αυτή η συγκεκριμένη τάση που ήδη έχει ε, προσδιοριστεί και αναφέρεται σε διεθνείς συζητήσει ε, για το θέμα της ασφάλειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με ευρυδικές λύσεις και απαντήσεις, ε, δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει την επένδυση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και σε ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών. Σε τέτοια καταστάσεις λοιπόν εμείς δίνουμε συμβουλές στην ε, κυβερνήσεις αλλά και στις αρμόδιους οργανισμούς να σκεφτούν αυτές τις συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να ελοπιθούν στο πλαίσιο της καταπολέμησης των υβριδικών απειλών κατά της ασφάλειας και να δοθούν τα κατάλληλα κονδύλια για να απαντηθούν αυτές οι απειλές. Ανάλογα δηλαδή με την αξιολόγηση των απειλών. Αυτά τα δύο θεματολόγια θα μπορούσε κάποιο να μιλήσει για μια μαλακή ατζέντα, παραδείγματο χάρη ε, προστασία τη κοινωνία των πολιτών, ε, των μέσων ενημέρωση, των υπερσπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της, ε, του σκληρού θεματολογίου. Τι συνδέονται. Εμεί θέλουμε να αξιολογηθεί και το επίπεδο τη δέσμευση δυνάμει τη αρχή ότι η επένδυση σε υβριδικέ απαντήσει θα πρέπει να είναι ανάλογη στο επίπεδο των υβριδικών απειλών. Είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσεις αν έχετε. Ευχαριστούμε κύριε Πομιανόφσκι, που μας παρουσιάσατε την ετήσια σας έκθεση και τις δραστηριότητες του Ταμείου. Έχουμε 10-15 λεπτάκια να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Να ευχαριστήσω και όσους ε, είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούνται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Ο κύριος Προνιού έχει το λόγο, πρώτος συνάδελφος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εκτελεστικό διευθυντή για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης. Με συγχωρείτε που δεν άκουσα το σύνολο της παρέμβασής σας. Όμως, τι λάβαμε την έκθεση, και την έχω μελετήσει προσεκτικά. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Καταρχήν συγχαρητήρια για το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία από το 2013. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον δεδομένων των στόχων που μπορεί να έχετε να ακούμε ή να διαβάζουμε ότι αποτελείται προστιθέμενη αξία προκειμένου να επιτρέψετε στη δημοκρατία στις χώρες ε, όπου δίνετε τις επιχορηγήσεις ε, να είναι καλύτερο το επίπεδο διαβίωσης. Στη σελίδα 15 βλέπω ότι το σχέδιο που σχετίζεται με τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, είναι πολύ μακριά σε σχέση με την υποστήριξη. Υπάρχει μια έκθεση που αφορά την πρόθεση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς, το χάρη. Πιστεύω ότι ίσω πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για αυτό το τελευταίο θέμα, δηλαδή την καταπολέμηση τη διαφθορά. Είτε μιλάμε ε, για την Ανατολική, την Νότια γειτονία μας, ε, αυτή η διαφθορά κάνει τους πολίτες ε, να αισθάνονται ότι δεν συμμετέχουν στα κοινά και υποσκάπτει την πολιτική και οικονομική εξέλιξη των χωρών αυτών. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε λοιπόν αυτό το παράγοντα. Δεύτερον, πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την Νότια Μεσόγειο οι περισσότερε πολιτικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωση, τα επόμενα έτη βρίσκονται στο νότιο τη Μεσογείου, καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, περιφερειακή σταθερότητα, απασχόληση των νέων ε, και χειρισμός, εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη, η ε, απαραίτητη δημοκρατική εξέλιξη για να απαντήσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και πέρα από το τι γίνεται στην Αλγερία έχουμε πολιτική ατονία και έχουμε όλο ένα και πιο χαμηλή συμμετοχή στι εκλογές σε όλες τις χώρες στην νότια όχθη της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν πώς η δική σας οργάνωση μπορεί να βελτιώσει τη δράση της στον τομέα αυτό και ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε σήμερα. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Ζιλ. Άλλα σχόλια από τους συναδέλφους. Όχι. Κύριε Πομιανόφσκι, θέλετε να απαντήσετε. Σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα ερώτηματά σας. Είναι απολύτως θεμητά και πολύ σημαντικά. Μιλώ και γαλλικά βέβαια, αλλά ε, συνήθως μιλώ στα αγγλικά γιατί τα γαλλικά μου δεν είναι τόσο πολύ καλά για να σας απαντήσω στα αγγλικά, γαλλικά κατευθείαν. You ask about, uh, specifically... Uh, Ρωτήσατε συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της διαφοράς στην uh, ανατολική γειτονιά της Ευρώπης. Είναι ουσιώδου σημασία στο κομμάτι αυτό, σε ό,τι αφορά τη στήριξη που δίνουμε στη Μολδαβία, στην Ουκρανία και άλλες χώρες. Και ταυτόχρονα είναι αλήθεια ότι είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι του πολιτικού ακτιβισμού γιατί γιατρεύει όλες τις ασθένειες. Προσπαθώντας αυτές οι χώρες να βγουν από το παρελθόν τους. Και επίση αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει και μια τρίτη διάσταση. Ένα τμήμα της διαφθοράς δεν είναι ε, παραδοσιακό, είναι και μεθοδολογία των μεγάλων γιντόνων να ε, ε, ελέγχουν την πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν και μεγάλοι εχθροί που, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε που είναι υπέρ του να διατηρηθεί η προτεραία κατάσταση. Επίσης, η, η, η ε, κοινωνία ε, εκτίθεται στην διαφθορά ε, κάθε μέρα, οπότε η κοινωνία είναι αυτή που πρέπει να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί. Και επίσης, είδαμε από πέρσι τεράστια ανάπτυξη φυσικών επιθέσεων σε ε, ακτιβιστές ε, που είναι αντίθετοι με τη διαφθορά. Κάποιους τους μαχαίρωσαν στην πλάτη και ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός ε, ε, ε έζησε. Έχουμε πάνω από 50 καταγεγραμμένες υποθέσεις. σε άλλους επιτέθηκαν στην Οδυσσό. Είναι λοιπόν πραγματικά αγώνας για τη ζωή για μερικούς ανθρώπους η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν είναι απλός ακτιβισμός, αλλά είναι πραγματικά αφοσιωμένοι στο στόχο αυτό. Και αυτή είναι η μόνη απάντηση που έχουμε. Πρέπει να το στηρίξουμε και αυτοί θα βρούνε τον τρόπο να μειώσουν την διαφθορά στη χώρα τους. Αλλά βεβαίως χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται προσπάθεια, όλη αυτή η διαδικασία και χρειάζεται και συντονισμένη προσπάθεια και από την διεθνή κοινότητα. Και εδώ και μιλώ για τα κρατικά κυρίως προγράμματα. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει πολιτική πίεση συνεχώς Σημαίνει αυτό να, ε, να προσπαθούμε να πιέσουμε τους ε, ηγέτες αυτών των χωρών ε, να βγουν από την καθιστική ατάξη τους και να αρχίσουν να ασχολούνται πιο, ενεργά και να στηρίζουν τους ανθρώπους που παλεύουν για την αντιμετώπιση της της διαφοράς. Μιλήσατε για πολύ συγκεκριμένε προτεραιότητες που έχουμε οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη δικές μας, όχι επειδή δεν θεωρούμε ότι είναι σημαντικές, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη και η σταθερότητα στην περιοχή είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά δική μας. Δεν είναι δουλειά δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία αυτό. Εμείς έχουμε πολύ περιορισμένα κονδύλια. Αυτό είναι θέμα γενικότερη πολιτική. Εμεί όταν ιδρυθήκαμε είχαμε ως δεδομένο ότι θα δημιουργήσουμε ένα πεδίο το οποίο θα συμπληρώνει τη δουλειά άλλων υπαρχόντων μέσων. Γι' αυτό εμείς επικεντρωνόμαστε στις δραστηριότητε που συμπληρώνουν τη μεγάλη εικόνα ας πούμε, και τα μεγάλα προγράμματα τα οποία ε, έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και μεγάλοι δωρητέ, διμερεί ή όχι. Εμεί επικεντρωνόμαστε στον ακτιβισμό των πολιτών, στα ανεξάρτητα ΜΜΕ, στου ε, νέου εισερχόμενου στην πολιτική σκηνή επίση, γιατί αυτά τα νέα πρόσωπα είναι πάρα πολύ σημαντικά ώστε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και να δώσουμε στου ανθρώπου μια αίσθηση ότι είναι δυνατό να υπάρξει αλλαγή. Υπάρχουν ε, νέα πρόσωπα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ήδη το έχουμε, έχουμε αποδείξει ότι φέρει προστιθέμενη αξία. Η δική μας η ε, μεθοδολογία είναι η προσέγγιση να είναι ευέλικτη, να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα και να συμπληρώσουμε τα πιο παραδοσιακά προγράμματα που ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν τα θέματα σταθερότητας στην περιοχή και ευημερίας ναι, άλλες φορές με καλά, άλλες φορές με αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό βέβαια δεν είναι ε, δική μου αρμοδιότητα να το σχολιάσω. Αλλά να πω κάτι για την Αίγυπτο. Εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει μια σημαντική εύκολη αντίφαση μεταξύ σταθερότητας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας της ε, κοινωνίας των πολιτών. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου, ο πρόεδρος Σίση, επιτίθεται και δημιουργεί ένα πάρα πολύ εχθρικό περιβάλλον προς την κοινωνία των πολιτών. Αν εξαφανιστεί η κοινωνία των πολιτών, όταν θα υπάρξει επανάσταση, όταν θα υπάρξει αναταραχή, γιατί κάποια στιγμή θα υπάρξει αυτή η στιγμή, γιατί η οικονομία της Αιγύπτου δεν πάει καλά, μόνο αυτή θα είναι η δύναμη που μπορεί να διατηρήσει την, και να προωθήσει την αλλαγή με έναν πολιτισμένο τρόπο. Αν εξαφανιστεί η κοινωνία των πολιτών, θα έχουμε μόνο ακραία φαινόμενα. Θα έχουμε μόνο ακραίες παρουσίες στην κοινωνία. Είτε αυτή θα είναι η ε, ε, κυβέρνηση, είτε θα είναι η ακραία ε, αντίπαλή της. Και άρα έτσι θα οδηγηθούμε σε άλλη μια καταστροφή με άλλους 200.000-300.000 πρόσφυγες στην Μεσόγειο προς την, να έρχονται προς την Ευρώπη. Οπότε το να, ευχα, το να επενδύουμε στην κοινωνία των πολιτών σημαίνει ότι επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη ευημερία, όχι μόνο στη βραχυπρόθεσμη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο από τους συναδέλφους. Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Και θα σας ξαναδούμε στην επόμενη έκθεση. Και τώρα... Παρόλο που προχωράμε καλά και έχουμε χρόνο στην διάθεσή μας, να αρχίσουμε με το επόμενο σημείο. Πάμε στο 6. Ενημέρωση από, για την ε, αποστολή της ΑΦΕΤ στη Σερβία και το Κωσοφοπέδιο, 27 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου. Εγώ ήμουν ε, ο πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας αυτής, οπότε να πω δύο λόγια. Και βεβαίως συνάδελφοι, ευχαρίστως να πάρετε το λόγο και να πείτε τη δική σας άποψη. Επικεφθήκαμε λοιπόν και τις δύο χώρες από τις 27 Φεβρουαρίου στις 2 Μαρτίου. Εγώ ήμουνα επικεφαλής της ε, επιστολής αυτής με άλλους πέντε ε, συναδέλφους. Νίνα Γκίλερ, Μαρμπρόκ, Ρίσαρτ Τσανέσκι, Ίγκο Σόλτες και Γιάρο Μιτσκόλιτσεκ. Ο στόχος του, του, της ε, επισκέψης μας ήταν να δούμε πώς έχει η πολιτική κατάσταση τόπου και να κάνουμε έναν απολογισμό της, ε, των σχέσεων ε, του Κωσόβου και τη Σερβία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τι γίνεται με τις συμπεφωνημένε μεταρρυθμίσει μεταξύ του διαλόγου που υπάρχει, για το διάλογο που υπάρχει μάλλον μεταξύ Βελγραδίου και Πρίστινα. Ε, κάναμε, περάσαμε μια μισή μέρα σε κάθε πόλη, στο Βελιγράδι και την Πρίστινα. Κάναμε συζητήσει ειλικρινή και ει βάθο με την πολιτική ηγεσία, με εκπροσώπου ε, και των, ε, των, ε, κυβερνητικών και των ε, κομμάτων τη αντιπολίτευση, με εκπροσώπου κοινωνία των πολιτών και με διπλωμάτε που βρίσκονται στη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Στη Σερβία εκφράσαμε την πλήρη στήριξή μα για την αφοσίωσή τη στον δρόμο τη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίσαμε βεβαίω ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη πρόοδο, κυρίω σε τομείς όπως το κράτο δικαίου και η ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Στο κοσυφοπαίδιο επαναλάβαμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει να κάνει με, την ε, στήριξη, με τη στήριξη για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και καλωσορίσαμε την πρόοδο που έχει γίνει στον ε, κλάδο ε, του, του κράτου δικαίου. Αλλά βεβαίω θυμίσαμε ότι η εφαρμογή όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι αυτή που θα καθορίσει και την επιτυχία του προγράμματο. Και στι δύο πόλει, και στο Βελιγράδι και στην Πρίστινα, Τονίσαμε την ανάγκη για να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δύο ε, πλευρών και ζητήσαμε και από, τις, από τα δύο μέρη να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα λύνει τα εκκρεμόντα θέματα πριν ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταστήσαμε απόλυτα σαφέ ότι και η Πρίστινα και το Βελιγράδι πρέπει να συμβάλλουν ώστε να υπάρξει ένα αγώγιμο περιβάλλον για να επιτευχθεί ο στόχο αυτό. Και οι αρχέ τη Πρίστινα θα πρέπει να ε, σταματήσουν τις, ε, ε, δασμού στα αγαθά 100% που παράγονται στη Σερβία και στη Βοσνία. Δεν θα σα εκπλήξει να σα πω ότι οι βασικοί μα συνομιλητέ στο Πρίστινα δεν πίστηκαν και δεν άλλαξαν γνώμη. Εμεί επαναλάβαμε τη θέση του Κοινοβουλίου στο να υπάρξει μια ε, συνολική νομικό δεσμευτική συμφωνία και η Σερβία και το κοσφοπέδο θα πρέπει να παραμείνουν πολυεθνοτικά και οποιαδήποτε ε, συμφωνία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή μόνο αν συμφωνηθεί και με, τους δύο, με τα δύο μέρη, συνάδει με την ε, διεθνή νομοθεσία και λαμβάνει υπόψη την συνολική σταθερότητα στην περιοχή. Πριν δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας, να ευχαριστήσω ε, τους ε, ε, όσους μας φιλοξένησαν στο βελγράδι και την Πρίστινα, τον πρέσβη, την, την πρέσβη, συγγνώμη, της, της Σερβίας, την κυρία Νατάλια Αποστόλοβα που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και τον εξοχότατο Σεμ Φαμπρίτσι, τον, τον πρέσβη στη Σερβία. και βεβαίω στι ομάδε του που μα έδωσαν πραγματικά μεγάλη στήριξη για την επίτευξη αυτή τη αποστολή. Και πριν και κατά τη διάρκεια και μα έδωσαν βεβαίω και επιτόπου πάρα πολύ καλέ συμβουλέ. Αυτά από μένα. Συνάδελφοι, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, σας ακούμε. Ο κύριος Κούλιτσεκ έχει το λόγο. Λοιπόν, ε, θέλω να να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπατε. Δεν υπάρχει και τσεχική διερμηνία. Θέλω να προσθέσω λοιπόν σε αυτά που είπατε ότι η επίσκεψη ε, μας έδωσε την ευκαιρία να έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ε, συναντήσεις με πολίτες ε, στο Βελιγράδι. Η κατάσταση στο Κόσοβο είναι πολύ διαφορετική, πολύ μακριά από την ε, Ευρώπη λόγω των ε, βίαιων συγκρούσεων ε, που έχουν γίνει στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Ο πρόεδρος ενημερώνει τον ομιλητή ότι υπάρχει τσεχική διερμηνία ο, ο κύριος Κόλτσεκ ε, λέει ότι μπορεί να μιλήσει και άλλες γλώσσες. Συνεχίζει όμως στα τσεχικά. Θα μιλήσω λοιπόν κύριε Πρόεδρε τσεχικά. Ναι, δεν υπάρχει συνήθως καμπίνα τσεχική, αλλά μιας και υπάρχει θα την αξιοποιήσω. Υπάρχουν λοιπόν στην, ε, στο Κόσοβο άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται ως πολιτικοί ενώ θα έπρεπε να είναι κατάδικοι για τα όσα έχουν κάνει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Κωσυφοπαίδιο είναι το ότι υπάρχει αδιαφάνεια όσον αφορά τα οικονομικά ε, στοιχεία και όπως ακούσαμε και από τον ε, Πολωνό συνάδελφο, τα πράγματα δεν ε, βελτιώνονται. Υπάρχουν ε, αμύθιτα ποσά που κυκλοφορούν στη χώρα, κατασκευάζονται νέοι δρόμοι, νέα, κτίρια, τεραστίων διαστάσεων και κανείς δεν γνωρίζει από ποιον και από πού έχουν χρηματοδοτηθεί αυτά. Σε ό,τι αφορά την Σερβία, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητήσει συγνώμη στη Σερβία για τη ζημιά που προκλήθηκε στη χώρα αυτή, στο περιβάλλον της χώρας αυτής, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Μια ζημιά ανυπολόγιστη με τη χρήση χημικών όπλων, τα οποία έχουν δηλητηριάσει το υπέδαφος της χώρας βομβαρδίστηκαν γέφυρες, δεκάδες. Μέχρι και σήμερα λοιπόν μπορεί κανείς να δει ότι η χώρα αυτή προσπαθεί να ξεπεράσει τις ε, σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες αυτών των βομβαρδισμών. Δεν ξέρω, δεν αναφερθήκατε σε αυτά, αλλά θα θυμάστε ότι ε, ε, και στις συναντήσεις μας οι αξιωματούχοι πολύ προσεκτικά ε, χειρίζονται και προσεγγίζουν αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτή τη χώρα γιατί εν μέρη ευθυνόμαστε και εμείς για τα όσα έχουν συμβεί εκεί. Επίσης, κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει είναι το, τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η παρουσία απεμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απομακρύνει κανείς από το υπέδαφος και από το περιβάλλον της χώρας. Οι δικέ μου εντυπώσει λοιπόν από την Σερβία, και δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που επισκέφτηκα το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη περιφέρεια της Ευρώπης, είχα επισκεφτεί τη χώρα αυτή ε, πολύ, πολύ συχνά όταν ήμουν ε, νέος. Αποτελεί λοιπόν αναπόσπαστο για εμένα τμήμα της Ευρώπης και νομίζω ότι η στάση μας απέναντι στη χώρα αυτή θα πρέπει να είναι θετική. Αυτά με δύο λόγια. Ελπίζω και στην επόμενη ε, θητεία να έχουμε την ευκαιρία να υπερβούμε τα προβλήματα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόλτσεκ. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο. Ε, Edward Κούκαρτ Κούκαν, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για την διμερή συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί δεν συμμετείχα στην αντιπροσωπεία. Μπορώ όμω να σα ε, πω δύο λόγια για αυτά που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ε, έγινε η κοινοβουλευτική ε, συνέντηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κούπστινα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ε, ήταν λίγο επίγουσα αυτή η συνάντηση γιατί τα πράγματα ήταν επιτακτικά. Καταφέραμε όμως να συζητήσουμε όλα τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική κατάσταση και τις σχέσεις μας με την Σερβία, τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας γενικώ. Υπήρχε λοιπόν καλή συμμετοχή και από τις δύο αντιπροσωπείες στη συνάντηση αυτή. και καλύψαμε όλα τα σημαντικά θέματα. Αναφέρθηκε δε και από τις δύο πλευρές ότι η Σερβία σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τις ε, προενταξιακές διαπραγματεύσεις και τονίστηκαν ε, ιδιαίτερα οι τομείς ε, στους οποίους υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται. Όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, για τρίτη συνεχή χρονιά στην ετήσια έκθεση η Κομισιόν αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόοδο στον τομέα αυτό και προφανώ είναι σημαντικό να σημειωθεί και να διαπιστωθεί πρόοδο και σε αυτό τον τομέα. Σε σχέση με τον ε, διάλογο ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα, οι συνάδελφοί μας από τη Σερβία μας εξήγησαν ποια είναι η δική του ε, οπτική θεωρούν ότι η μεταχείριση που τους επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δίκαιη, ακριβώς διότι δεν ευθύνονται εκείνοι για, την, για το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει ο διάλογος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διαδραματίσουμε ένα πολύ ενεργότερο ρόλο, γιατί ε, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Και οι δύο πλευρές θα περιμένουν μια όθηση από εμάς αν θέλετε προκειμένου να ξαναξεκινήσει ο διάλογος και να ξεπεραστεί η κρίση που υπάρχει. Ε, αναφερθήκατε και εσείς κύριε Πρόεδρε στην αύξηση των δασμών. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων καταφέραμε να εγκρίνουμε την κοινή διακήρυξη που υπεγράφει Θεωρώ γενικά ότι η συνάντηση αυτή ε, ήταν θετική, στέφθηκε με επιτυχία και εκφράστηκε η ελπίδα ότι το νέο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο θα συνεχίσει το θετικό έργο που επιτελέστηκε από τα τωρινά μέλη της αντιπροσωπείας μας. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν για τις πρόσθετες αυτές παρατηρήσεις σε σχέση με την ε, συνάντηση που έγινε την ε, προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, η οποία ήταν ε, σύντομη αλλά και πολύ έντονη. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Ωραία. Αυτή ήταν η ενημέρωση λοιπόν σε σχέση με την αποστολή της ε, Επιτροπής ΑΦΕΤ στη Σερβία και στο Κωσυφοπαίδιο και περνάμε στο σημείο 7, αποστολή της ΑΦΕΤ στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Κάναμε λοιπόν μια επίσκεψη και σε αυτές τις δύο χώρες για να πάρουν το πράσινο φάνο για να ξεκινήσουν ε, οι πρωταξιακές συνομιλίες ε, φέτος ε, τον Ιούνιο. Είχαμε μία αποστολή επτά μελών υπό την ηγεσία του κυρίου Κέλλαν που συνάντησε άτομα από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Έλαβε χωρί επίσκεψη στα μέσα μια πολιτική κρίση στην Αλβανία με την αντιπολίτευση να αρνείται η κοινοβουλευτική της ε, θητεία στη Βορεια Μακεδονία. Ε, είχαμε την επίσκεψη κατόπιν της επικύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσφών και εν ώψη της προκλοκής εκστρατείας για τις εκλογές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξοχότατους ε, Σάμιλ Μπόργκερ, τον πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βορεια Μακεδονία και τον κύριο Λουίτζι Σορέκα, τον πρεσβευτή στην Αλβανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ομάδες τους για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω και τους οικοδησπότες μας στα Τύρανα και στην και στα Σκόπια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Τούνε Κέλαμ, αν ήταν εδώ. Δυστυχώ απουσιάζει. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Κούκαν. Για τη Βόρεια Μακεδονία. Παρακαλώ, πάρτε το λόγο, ναι. Εγώ συμμετείχα ως μέλος της αντιπροσωπείας ε, στη επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία και μας ε, ενθάρρυναν να, ε, να υλοποιήσουμε εκεί συνεδριάσεις και συνομιλίες. Επίσης είχαμε και μία συνάντηση με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Ε, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική συνάντηση αυτή, γιατί ε, η κατάσταση είναι ότι θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό ΖΑΕΦ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί συνεχίζεται ο πολιτικός διάλογος σε ψηλό επίπεδο και συμφώνησαν να συμμετέχει και η αντιπολίτευση στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Δημιούργησαν δύο ομάδες εργασίας με την πλήρη συμμετοχή της αντιπολίτευσης και αυτό σημαίνει ότι αν και η αντιπολίτευση δεν υποστήριζε τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως ε, λένε, θεωρούν ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό και τα δύο μέρη τώρα επικεντρώνονται στις ε, εκλογές, τις προεδρικές, που θα λάβουν χώρα αργότερα τον Απρίλιο. Όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να είναι διαφανείς και δίκαιες οι εκλογές αυτές. Έτσι, λοιπόν, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος ε, στις εξελίξεις ε, στη Βόρεια Μακεδονία και θα ενισχυθεί αυτή η πρόοδος. Έτσι, λοιπόν, μπορέσαμε να συναντήσουμε όλους τους ηγέτες και η συζήτηση με αυτούς ε, ήταν πολύ θετική και νομίζω ότι πρέπει να τους υποστηρίξουμε στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις φιλοδοξίες της Βόρειας Μακεδονίας ε, για να λάβει την ημερομηνία για την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Λόγω των ε, θετικών πολιτικών αλλαγών που είναι ορατές πρόσφατα, αυτό θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του Συμβουλίου. Και νομίζω ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια τέτοια εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έντουαρτ, για τα σχόλιά σου, για την κατάσταση για τη Μακεδονία. Περαιτέρω σχόλια υπάρχουν, όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως, εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωση για τις δύο αποστολέ στα Δυτικά Βαλκάνια. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εκθέσεις αποσπολής ε, στο ιστοσελίδα της ΑΦΕΤ, ε, στο τμήμα Notice to Members. Ε, τώρα, θα δούμε πότε θα θετηθούν, θα 29η έκθεση πρόοδου. έκθεση πρόοδου. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου. Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια ακόμη συνεδρία της Επιτροπή ΑΦΕΤ λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές γιατί μιλήσαμε με την ομάδα του Επιτρόπου Χάν και θέλουμε να έχουμε πληροφορίες από πρώτο χέρι σε σχέση με το περιεχόμενο της νέας έκθεσης πρόοδου. Πριν να ενημερωθούν ε, φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, αλλά προσθέ... σκοπεύουμε να έχουμε πρόσθετη συνεδρία στις 29 Μαΐου. Τώρα, είμαστε 35 λεπτά μπροστά στο χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Πολύ ωραία. Σημείο 8. Πρόληψη των συγκρούσεων και διαμεσολάβηση. Υφιστάμενη ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μελλοντικέ προοπτικέ. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Μονάδα Διαμεσολάβηση Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ε, Πού θέλουν να καθίσουν συγκεκριμένοι, θέλουν να έρθουν εδώ στο πάνελ. Σα καλώ να έρθετε εδώ, στο Προεδρείο. So. Κυρίε και κύριοι, περνάμε στο σημείο 8. Και καθώ προσεγγίζουμε το τέλο αυτή τη θητεία και πρόσφατα υιοθετήσαμε τι εκθέσει για την οικοδόμηση των Ευρωπαϊκών Ικανοτήτων για την πρόληψη και τη διαμεσολάβηση των σειράξεων και το ρόλο και το παιδί εφαρμογή των ειδικών προσώπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καιρό να συζητήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε βάση τη κληρονομιά που έχουμε από αυτή τη θητεία και των επιτευγμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε για μια συνολική προσέγγιση, συνδυάζοντα την ασφάλεια, τη διπλωματία και την ανάπτυξη και για πιο ισχυρό πολιτικό και θεσμικό συντονισμό εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο έχει έναν εξέχοντα ρόλο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και για τη δημοσιολάβηση και για το διάλογο. Ο συνάδελφο, ο κ. Κούκαν, ο οποίο είναι ένα από σε επικεφαλή στον τομέα αυτό θα μα πει περισσότερα για την πολιτική διαμεσολάβηση του Κοινοβουλίου και για το διάλογο. Κατόπιν ο κύριος Μάικλ Κίτινγκ, τον οποίο καλωσορίζω ένθερμα, εκτελεστικό διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη, θα παρουσιάσει τι δραστηριότητε και τη στρατηγική του Ινστιτούτου σε ό,τι αφορά την επίλυση των σειράξεων και την ειρήνευση. Και τέλος, ο κύριος Ρενέ Φανές, ο οποίος από ό,τι με έρχεται, είναι ο επικεφαλής του τμήματος για την πρόληψη των συγκρούσεων και την υποστήριξη διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Κούκαν, ο οποίος ήταν ε, ενεργός στην υποστηρίξη την ε, δημιουργία του Ινστιτούτου, το οποίο ταιριάζει γιορτάζει τώρα την πέμπτη επέτειο. Θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Κούκαρ για 10 λεπτά και κατόπιν ο κύριος Κίτιν και μετά ο κύριος Φανές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την χρονική στιγμή που οργανώσατε αυτή την συνάντηση, γιατί είναι δύο εβδομάδες μετά την υιοθέτηση της έκθεσης για την επίλυση σειράξεων και τη διαμεσολάβηση. Και επίσης είναι και η πέμπτη επέτειος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ειρήνης. Είναι μια στιγμή λοιπόν να ξανασκεφτούμε την το τι αφήνει πίσω το, το κοινοβούλιο και τι περιμένει το νέο, τους νέους ευρωβουλευτές και τους νέους επιτρόπους. Να μην ξεχνούμε ότι όταν μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση σειράξεων και στη διαμεσολάβηση, μπορούμε να απαντήσουμε συνεκτικά στους πολίτες μας και στο ευρωβαρόμετρο, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ενεργός στις εξωτερικές σχέσεις για να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα και να μπορεί να επιφέρει ειρήνη σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα υπογράμμιζε την ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική ε, αντιμετώπιση σειράξεων και τα αντίστοιχα εργαλεία και να υποστηρίζονται όλες αυτές οι διαδικασίες μέσω της διαμεσολάβησης. Πρόσφατα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα ε, μίλησαν ε, για σημαντικά, με σημαντικά επιχειρήματα από οικονομική πλευρά για την διαμεσολάβηση και για την αντιμετώπιση σειράξεων, έτσι ώστε να δούμε το κόστος και το όφελος της, ε, των σχετικών στρατηγικών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε βίαιες σειράξεις. Κάποιες από τις πιο μακροχρόνιες σειράξεις ε, που περιλαμβάνονται και στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και στη γειτονιά μας, χρειάζονται μεγαλύτερη πολιτική παρέμβαση μέσω ενίσχυσης της διαμεσολάβησης για να επιφέρουμε σταθερότητα, να μειώσουμε τη μετανάστευση και να παράσχουμε οικονομική ανάπτυξη για τους ε, γείτονες και τους πολίτες μας. Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει μια πολύ καλή γενική εικόνα για το τι, ε, τι μέσα αντιμετώπισης των σειράξεων υπάρχουν ήδη σε όλα τα, μέσα από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και επίσης ε, προτείνει και κάποιες καινοτόμες ιδέες για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, τρο, με τρόπο αποτελεσματικό προς το κόστος. Επίσης ε, λέει, δείχνει η έκθεση πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γίνει νέος παίκτη σε αυτή τη σκακέρα με την δική του ξεχωριστή ε, παρέμβαση στην, μέσω της πολιτικής κοινοβουλευτικής διαμεσολάβησης. Μπορώ να πω από την εμπειρία μου ότι η συνεργασία με τους ε, ε, αξιότιμους συναδέλφους Βάινερ και Φλέκενστάιν και με τον Επίτροπο Χάν στην ε, Βόρεια Μακεδονία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική όταν όλα τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη-μέλη της συνεργάζονται. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλάμβανε και βασίστηκε σε μια ιδέα που ήδη έχει εφαρμοστεί από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου ζητείται υψηλού επίπεδου διαβούλευση και ένα αντίστοιχο συμβουλευτικό όργανο με συμπερίληψη και με νυν και παλαιών ε, ευρωβουλευτών. Υπάρχει μια πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση που δεν θα κοστίσει πολύ, αλλά θα συνδυάσει τα πολιτικά δυνατά μας στοιχεία. Να προσθέσω τώρα δύο πράγματα σε σχέση με τη δική μου εμπειρία, τώρα που είναι το τέλος της θητείας. Το 2015 ο Επίτροπος Χάν ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει να στηριχθούν οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η πολιτική κρίση στην πρώην Ιουγκοσλαβική ε, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απήντησε θετικά και δημιούργησε την διαμεσολαβητική ομάδα τριών ευρωβουλευτών με τον κύριο Φλέκενστάιν, τον κύριο Βάγγελ και εμού. Και τα τρία αυτά χρόνια δουλέψαμε ως ομάδα με τον Επίτροπο Χάν. Καμιά φορά ε, δουλεύαμε από κοινού και με τα Σκόπια. Προσπαθήσαμε να ε, ε, συντονίζουμε τις συναντήσεις μας με τον Επίτροπο ώστε να έχουμε ε, το, μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο μόχλευσης. Αλλά πάντα δουλεύαμε ως ευρωπαϊκή ομάδα και είχαμε πάντα όλοι τον ίδιο στόχο. Να συνεργαστούμε με τα πολιτικά κόμματα για να βοηθήσουμε τη χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση στην οποία βρίσκεται. Διαθεσμικά δουλεύοντας ε, μπορέσαμε να έχουμε τη βοήθεια και τον, ε, την, ε, την, της Γενικής Διεύθυνσης, της ομάδας της διαμεσολάβησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων και τον πρέσβη Σβόγκαρ αλλά και τον πρώην πρέσβη Άιβο Όγκαρ. Ήταν πραγματικά πολύ αποτελεσματική η παρέμβαση και η δουλειά όλων. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε περήφανοι γιατί αυτή η πρώτη ε, πρωτοβουλία διαμεσολάβησης ε, επέτυχε σημαντικά αποτελέσματα για να υποστηρίξει τη χώρα, χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσε η χώρα αυτή να έχει κάνει ε, την σημαντική αυτή αλλαγή, να πει το ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να γίνει μέλος και να υιοθετήσει το νέο όνομα της Βορειού Μακεδονίας. Συνεχίζουμε την υποστήριξη στην χώρα αυτή για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά προς το παρόν δεν τονίζουμε τον ρόλο της διαμεσολαβητικής ομάδας. Αυτό που τονίζουμε τώρα είναι η στήριξη προς το διάλογο μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια πολιτική νοοτροπία διαλόγου και συμβιβασμού, που θα τους ε, βοηθήσει, θα βοηθήσει την εθνική τους ε, αντίσταση ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, να προλάβουν μελλοντικέ ε, κρίσεις. Ίσως αυτό να είναι απλό ή να σας φαίνεται απλό, αλλά για κάποιες χώρες στη Δυτικά Βαλκάνια βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουν το θέμα του συμβιβασμού και τους παίρνει πολύ χρόνο για να το πραγματοποιήσουν. προσπαθούμε να προχωρήσουμε, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο στόχο. Ε, επικεντρωνόμαστε λοιπόν στο να καλλιεργήσουμε αυτές τις δραστηριότητε έτσι ώστε να ε, τα καταφέρουμε, γιατί πραγματικά είναι επίγουσα ανάγκη. Ο διάλογο για να υποστηριχθεί και ο διακομματικό ε, διάλογο γίνεται ω εξή. Υπάρχουν νέε δυνατότητε μέσω ας πούμε, του διαλόγου Ζαμονέ που έχει εδραιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί μια ειδική μεθοδολογία διαμεσολάβησης και ενισχύει τις Δραστηριότητε βεβαίως του οίκου του Ζαμονέ έξω από το Παρίσι. Υπάρχει χώρος για διάλογο μακριά από τα φώτα των Βρυξελών και ο διάλογο Ζαμονέ χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ουκρανία με την ε, μεγάλη επιτυχία ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των ε, ε, κομμάτων στην Ουκρανία. Ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ και ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Κόξ, ήταν επικεφαλής της διαδικασίας αυτής και ήταν πραγματικά ε, είχαν ηγετικό ρόλο στη μεθοδολογία Ζαν Μονέ και στο, στην εφαρμογή του μέσου Ζαν Μονέ. Η της εργασία του Ζαν Μονέ ήταν ρεαλιστική, συγκεκριμένη και, ε, και μιλούσε για ε, επικεντρωμένο διάλογο που επιτυχάνει την ομοφωνία έτσι ώστε να προωθηθούν όλες οι δραστηριότητες διαλόγου Ζαν Μονέ. Τώρα χρησιμοποιούμε την ίδια μεθοδολογία για τα πολιτικά κόμματα στη Βόρειο Μακεδονία. Και ο διάλογος αυτός γίνεται στη χώρα. Ήταν η δική τους επιθυμία. Δεδομένων και των θετικών εξελίξεων λοιπόν των, α, της όλης ιδέας του διαλόγου Ζαμονέ, ο Επίτροπος Χάν προσφάτως μας ζήτησε να διευρύνουμε το μέσο αυτό πέραν της Βορείου για να καλύψει όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό το σημείο επίσης ε, στηρίχθηκε και από την έκθεση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια πριν από δύο εβδομάδες. Από την εμπειρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια σημεία. Ένα είναι η άμεση ανάγκη για συντονισμένη πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Η στενή διαθεσμική συνεργασία δείχνει μέσω της κοινή αυτής προσέγγισης που ξεκίνησε ο Επίτροπος Χαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και τον, και τον πρέσβη στα Σκόπια ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Η στενή συνεργασία σε επίπεδο υπηρεσιών επιτρέπει ε, καλύτερη στήριξη και τέλος τον, έχω τονίσει πολλές φορές τον πολιτικό ρόλο που έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργώντας περισσότερες μικτές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση σειράξεων και τη διαμεσολάβηση. Γιατί Όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Παγκόσμια Τράπεζα έχουν πει επανειλημμένω, η αποτελεσματική ε, διαμεσολάβηση και από πλευρά αποτελέσματο και, χρο... και κόστους σημαίνει κυρίω την πολιτική βούληση για να δράσει κανεί. Και αυτό υπογραμμίζεται από, το συντονισμένο... από τη συντονισμένη στήριξη μέσω των θεσμικών οργάνων που ε, είμαι πολύ ικανοποιημένο που μπορώ να σα πω ότι έχουμε δείξει επανειλημμένω μέσω τη ομάδα και αναφέρεται και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι μπορούν να το υποστηρίξουν και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ειρήνη, αλλά και οι συνάδελφοί σα. Η αντιμετώπιση σειράξεων μπορεί να είναι δύσκολη χωρίς να, αν, όταν δεν παρεμβαίνουν οι απόψεις των κρατών μελών, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση μέσω των θεσμικών οργάνων. Αυτό αντικατοπτρίζει και την πραγματικότητα πρέπει να έχουμε μόνο ένα ρόλο να παίξουμε και για να επιτύχουμε το στόχο μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε και όλες τις δυνατότητες μόχλευσης μέσω όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Edward Κούκαν, πάντοτε πολύ εύστοχος. Να δώσω το λίγο στον Μάικλ Κίτινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μικρόφωνο του μιλητή σας παρακαλούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τον ρόλο της ΑΦΕΤ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το γεγονός ότι συνέβαλε σημαντικά στη θέσπιση ε, αυτού του προγράμματος. Εγώ, ξέρετε, ε, σχετικά πρόσφατα ήρθα στις Βρυξέλλες, ήμουν ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Σομαλία και είναι μεγάλη μου τιμή που μου δόθηκε η δυνατότητα να τεθώ επικεφαλής αυτού του Ινστιτούτου, αυτού του οργάνου. Γνωρίζετε ε, κάποιοι ότι το EIP ε, δημιουργήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Ευρώπης όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων, την επίλυση διαφορών, τον διάλογο και τη διαμεσολάβηση. Επί της ουσίας λοιπόν επιτελούμε αυτό το έργο με τρεις τρόπους. Θέλω όμως να τονίσω ότι η δοντολογική μας ε, κατεύθυνση είναι πάντοτε να έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας ε, τα συμφέροντα των ανθρώπων που πλήττονται από τις συγκρούσεις, τη βία ή που κινδυνεύουν από τις συγκρούσεις και τη βία όπου και αν βρίσκονται, είτε βρίσκονται σε εύθραυστες, εύθραυστες χώρες είτε στην Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από πέντε χρόνια όταν δημιουργήθηκε το EIP δεν νομίζω ότι οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης ήταν όσο έντονες όσο είναι σήμερα. Οι τρεις τομείς λοιπόν στους οποίους εργαζόμαστε είναι η πολιτική, η πράξη και οι εταιρικέ σχέσεις ή καλύτερα να το πω πλατφόρμες για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων. Όσον αφορά την πολιτική, ε, κάνουμε αυτά στα οποία αναφέρθηκε και ο προηγούμενος ομιλητής. Δηλαδή, κατάρτιση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων από ευρωπαϊκούς φορείς για την εμπλοκή τους και τη συμμετοχή τους σε εύθραυστες χώρες, όπως είναι στον τομέα της πρόληψης των συγκρούσεων, της επίλυσης συγκρούσεων. Για παράδειγμα, οργανώνουμε διακριτικές συναντήσεις για συγκεκριμένες χώρες, για συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά δεν λειτουργούμε ω ε, δεξαμενή σκέψη, αν και δεν υποτιμούμε καθόλου κάτι τέτοιο, αλλά προσπαθούμε πάντοτε να προσδιορίσουμε πράγματα που πραγματικά μπορούν να γίνουν, απτές ενέργειες δηλαδή. Μια, ένα είδο δραστηριοποίηση και συμμετοχή που μπορεί να ενθαρρύνει το διάλογο, να μειώσει τη βία και να διευκολύνει τι ειρηνευτικέ διαδικασίε. Και η ανάγκη για τέτοιου είδου παρεμβάσει είναι τεράστιε. Εγώ ε, πριν από λίγες μέρες ε, γύρισα από το Αφγανιστάν, όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο της χώρας, τον επικεφαλής ε, του Συμβουλίου Ειρήνης, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματίες, γυναίκες και πραγματικά εκφράζονται τεράστιες ανησυχίες για το πώ οι συζητήσει για το μέλλον τη χώρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Και θεωρώ ότι ο δικό μα ρόλο στη συνεργασία μα με του Ευρωπαίου εταίρους μα, με τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα αυτή, είναι ε, το να καθορίσουμε ποια θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία και μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Αυτά όσον αφορά τον τομέα της πολιτικής. Στην πράξη ε, δραστηριοποιούμαστε σε 12 χώρες ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε με εταίρους για πολύ απτές δράσεις. Όπως για παράδειγμα στην Ιεμένη, όπου διευκολύνουμε τον ε, διάλογο μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών με απότερο στόχο τη συμφιλίωση των δύο πλευρών. Εργαζόμαστε στη Συρία όσον αφορά τον ασφαλή επαναπατρισμό των προσφύγων Μιλάμε, ε, δραστηριοποιούμαστε στο κέρας της Αφρικής για την πρόληψη του βιοεξτρεμισμού. Βοηθούμε μια σειρά από χώρες να ενισχύσουν τους δικούς τους μηχανισμούς και ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών. Αυτά όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι. Όσον αφορά τις εταιρικέ σχέσεις μας, θέλουμε να τις διευρύνουμε και να διευρύνουμε την πλατφόρμα εκείνων των φορέων που μπορούν να συμβάλλουν θετικά και ενεργά στην επίλυση διαφορών και την πρόληψη συγκρούσεων. Και σε αυτό βεβαίως εντάσσονται ε, ω αναπόσπαστο τμήμα οι βουλευτέ, ευρωβουλευτέ και εθνικοί βουλευτές. Και βεβαίως ε, μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να συμπεριλάβει τους επιχειρηματίες, τους ε, επαγγελματίες της ασφάλειας. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το, η, το, το ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την, για την Ειρήνη. Γιατί ένα από τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει είναι ότι δεν μπορεί να επιληθεί μια σύγκρουση χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που αναφέρατε και εσείς. Αυτή η ήπια ε, προσέγγιση είναι εξίσου σημαντική με την σκληρή προσέγγιση. Ακόμη και ε, στην οικοδόμηση και την κατασκευή ειρηνευτικών μηχανισμών και Δεν αρκεί να έχει μια χώρα μυστικές υπηρεσίες, στρατό και αστυνομία. Χρειάζεται να υπάρχει και μια οικοδόμηση θεσμών, κρατικών, που θα διευκολύνουν την ε, διατήρηση της ειρήνης. Και αυτή θα πρέπει να είναι η προοπτική μας. Και όχι μόνο να δίνουμε την προσοχή μας σε ε, αξιωματούχους επαγγελματίες της ασφάλειας, στο στρατό και την αστυνομία. Είναι εξίσου σημαντικά και τα άλλα. Γι' αυτό και θέλουμε να διευρύνουμε τους φορείς που συμμετέχουν στις πλατφόρμες μας. Όσον αφορά την ε, συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρούμε ότι η ΑΦΕΤ είχε μια ε, τεράστια συμβολή και θα έχει στο μέλλον μια τεράστια συμβολή στο να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων και θα συντονιστεί και θα συνδυαστεί η πολιτική και η οικονομική στήριξη σε εκείνους που τη χρειάζονται και που την αξίζουν, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς μέσω της ε, παρέμβασής μας σε εύθραυστες χώρες, στη γειτονία της αλλά και πέραν αυτής, προκειμένου να ε, προληφθούν οι συγκρούσεις. Διότι το αντίθετο, η αποτυχία στο να προληφθούν συγκρούσεις θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την Ευρώπη όσον αφορά τον εκτοπισμό, την ε, επισφάλεια και τις απρόβλεπτε πολιτικέ συνέπειε που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια αποτυχία. Χαιρετίζουμε την πολύ φιλόδοξη προσέγγιση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την πρόληψη συγκρούσεων και την ειρηνευτική διαδικασία και πρέπει να πω ότι κάποιε από τι προτάσει σα είναι πολύ ενδιαφέρουσε και πολύ καινοτόμε και θέλουμε κύριε Πρόεδρε να έχουμε συνεργασία μαζί σα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιε από τι ιδέε σα. Επίσης, με διάφορους τρόπους ε, συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Υπάρχει ένας αριθμός ε, ευρωβουλευτών, ε, ευρωβουλευτών που έρχονται σε εμάς ως παρατηρητές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έχει βοηθήσει σε κάποιες δραστηριότητες διαμεσολάβησης, μέσω της κατάρτισης που έχει παράσχει σε αξιωματούχους. Θέλουμε αυτές οι διαδικασίες να, διευρου, να διευρυθούν προκειμένου να πολλαπλασιαστούν και οι επιλογές που έχουμε για την επίτευξη των ε, ειρηνευτικών διαδικασιών. Θέλω όμως να πω κύριε Πρόεδρο ότι όταν συζητάτε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή ή η προσήλωση στο, στην, στον πολυμερή χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων οι γυναίκες, ο τομέας ε, της πρόληψης συγκρούσεων και της ασφάλειας. Υπάρχει πάντοτε αυτή η διάσταση της πρόληψης και της διαμεσολάβησης και δεν θέλω να σας καλέσω μάλλον να το λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας αυτό γιατί οι επιπτώσεις των συγκρούσεων είναι τεράστιες και νομίζω ότι δεν είμαστε αρκετά ε, ανθεκτικοί ε, ε, όσον αφορά ε, την προετοιμασία την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πρόληψη των συγκρούσεων και με χαρά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με ευρωπαϊκά κράτη που ε, είναι τόσο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα κράτη της Ευρώπης τα οποία έχουν μεγάλη συμβολή στην πρόληψη συγκρούσεων, Νορβηγία, Ελβετία που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλα αυτά έχουν πολλά να προσφέρουν. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ειδικό της βάρος, τις αξίες της, το διπλωματικό της δίκτυο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες, σε συγκεκριμένα ζητήματα, μια συμβολή η οποία θα ενισχύσει τον ρόλο της Υπήρου. Σας ε, θέλω λοιπόν να ε, σταματήσω εγώ λίγο νωρίτερα από ότι ο προηγούμενος ομιλητής, 34 ε, δευτερόλεπτα ακριβώς. Μάλιστα, 24 δευτερόλεπτα, έναντι 21. Πολύ καλά. Κύριος Φανές έχει φτάσει, εν μεταξύ αρχίσαμε λίγο νωρίτερα και μπορώ να σας δώσω κατευθείαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τον Μάικλ και αναφέρα μία σειρά εταίρων. Και είμαι σίγουρο ότι δεν άφησε σκόπιμα την υπηρεσία εξωτερικής δράσης εκτός του καταλόγου. Πολύ ωραία. Καταρχήν, να αναγνωρίσω τη σημασία της έκθεσης και του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σημασία της πρόληψης των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Και θέλω να συγχαρώ την ΑΦΕΤ ε, για την έκθεση αυτή και όσου συμμετείχαν στην εκπονησή τη. Πραγματικά ακολουθεί το σκεπτικό που είχαμε και εμείς, δίνει έμφαση στην εξάλληψη των αιτιών των σειράξεων και προωθώντας ε, ε, μεταρρυθμίσεις και το να θέσουμε την ανθρώπινη ασφάλεια στο επίκεντρο των δρασιών μας. Θα ήθελα να σας πω πώς εμείς βλέπουμε την πρόληψη των συγκρούσεων. Πέρσι τον Ιούνιο εκπονήσαμε μία έκθεση που λέγεται «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ω Παγκόσμιο Παίκτη για την πρόληψη των συγκρούσεων». Το συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη και σε λίγες γραμμές παρουσιάζει τις κύριες διαστάσεις της προσέγγισης ε, της ΕΕΔ για την πρόληψη των συγκρούσεων. Η βασική αρχή που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι η πρόληψη των σειράξεων απαιτεί στο να εργαζόμαστε σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Ε, κανένας ε, δεν μπορεί μόνος του να αποτρέψει μια σύραξη, κανένα μέσο δεν μπορεί να το πράξει από μόνο του. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι πρέπει όλα τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα συνενώσουμε για να δημιουργήσουμε συνέργειες και να εργαστούμε σε όλα τα διάφορα επίπεδα και τα στάδια μιας ε, σύραξης. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ και να σας πω με δύο λόγια την ε, αναδιοργάνωση που είχαμε εντό τη υπηρεσία εσωτερική δράση. Ίσως κάποιοι γνωρίζετε τι συνέβη στο παρελθόν. Είχαμε ένα τμήμα ε, που Ε, πρίζων ε, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει αυτό το ακρονίμιο. Έτσι λοιπόν ε, το πρίζων ως τμήμα έχει γίνει τώρα διεύθυνση. Έχουμε τώρα μια πλήρη διεύθυνση που περιλαμβάνει μια σειρά άλλων υπηρεσιών και ο στόχος αυτής της αναδιάρθρωσης είναι ότι θεσμικοποιήσαμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το η νέα διεύθυνση λοιπόν φέρει το όνομα ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια και την ειρήνη. Συμμετέχουν 89 ε, άτομα σε αυτή τη διεύθυνση και φυσικά θα έχουμε τις περισσότερες ικανότητες να προωθήσουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω τώρα στην πρόληψη των συγκρούσεων. Η πρώτη διάσταση, τέσσερις είναι συνολικά, είναι λοιπόν η πρώτη ότι αν ε, θέλουμε σοβαρά να προλάβουμε τις συγκρούσεις ε, θα πρέπει να καθοδηγήσει στην πολιτική προσοχή. Νομίζω ότι είστε τελευταίοι στου οποίου πρέπει να εξηγήσω πόσο σημαντική είναι η πολιτική προσοχή. Θα πρέπει να αυξήσουμε λοιπόν την πολιτική προσοχή για την πρόληψη των σειράξεων. Το δεύτερο που χρειαζόμαστε είναι τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία και έχουμε αρκετά. Και νομίζω ότι έχουμε βάλει πολύ μεγάλε προσπάθειε στο να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων. Θα αναφέρω τρία. Το πρώτο είναι το σύστημα εγκύρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλει κάποιος να προλάβει μια σύγκρουση, ποιες συγκρούσεις ε, θα προλάβεις, ποιες χώρες είναι σε κίνδυνο ξεσπάσει μια σύγκρουση, μια σύραξη, πώς το ξέρεις. Έχουμε λοιπόν έχουμε ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για τις σειράξεις. Και αυτό μας δίνει μια ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Μας ενημερώνει για τις χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο να υπάρξει μια βίαιη σύγκρουση. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Η κοινή ε, ανάλυση σειράξεων φυσικά γίνεται ε, με έναν τρόπο που λαμβάνει υπόψη και τα φύλλα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και μα οδηγεί στην ολοκληρωμένη προσέγγιση. Γιατί αν δούμε μια σύραξη με τον ίδιο τρόπο και συμφωνήσει ε, με του παράγοντε που οδηγούν στην ξέσπαση τη σύραξη, τότε μπορεί να καταλήξει και σε μια συντονισμένη προσέγγιση για το πώ να προχωρήσει. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι ότι πρέπει να έχεις την ικανότητα να προσλάβει εμπειρογνώμονε ε, τελευταία στιγμή για να αναπτυχθούν επιτόπου. Θα πρέπει να έχεις λοιπόν πόρους και έχουμε μια σύμβαση πλαίσιο χάρη σε εσά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πριν ε, δύο χρόνια δημιούργησε αυτό το χώρο που έχουμε στον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούμε να προσλάβουμε εμπειρογνώμονες ε, την τελευταία στιγμή και καθημερινά αυτό το εκτιμούμε. Και φυσικά επίση πρέπει να έχει, και παίρνω στο τρίτο, πρέπει να ενδυναμώσει τι εσωτερικέ σου ικανότητε. Πρέπει να έχει ανθρώπου με του οποίου να μπορεί να συνομιλήσει. Πρέπει να έχει συναδέλφου εντό τη υπηρεσία εξωτερική δράση και εντό κομισιών για να συνομιλήσει μαζί του για το θέμα τη πρόληψη των συγκρούσεων. Ε, πρέπει να έχει ε, μια κοινή γλώσσα. Δεν αρκεί να υπάρχει ένα τμήμα ε, που θα καθοδηγεί αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ε, την ε, μαθήματα κατάρτισης ε, και στην υπηρεσία εξωτερική δράση, αλλά και στο τότε της Κομισιόν για κάποια θέματα βασικά και εργαζόμαστε τώρα για τη δημιουργία μιας κοινότητας ατόμων που ασχολούνται με το θέμα αυτό στην πράξη. Και το τελευταίο είναι οι εταιρικέ σχέσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνη τη να τα καταφέρει. Πρέπει να συνεργαστούμε με του εταίρου μα και να πτήσουμε πολύ ε, σημαντικέ συμπράξει με τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε το διάλογο με τα Ηνωμένα Έθνη που λαμβάνει χώρα σε τη βάση. Και Επίσης, οικοδομούμε παρόμοιες σχέσεις ε, με τον ΟΑΣΕ. Έχουμε και εκεί σημαντικέ ανταλλαγές απόψεων και με την Αφρικανική Ένωση. Τώρα, αν δούμε το μέλλον, αν θέλουμε να, αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς, πρέπει να υπάρχουν πόροι. Και αναφέρεται ορθά η έκθεση στην ανάγκη να έχουμε επαρκείς οικονομικούς πόρους. Για μένα αυτό είναι ένας από τους τομείς όπου πρέπει να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο μελλοντικό, θα έχουμε επαρκείς πόρους που θα έχουν κατανεμηθεί για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Νομίζω ότι έχω αρκετό χρόνο να σας αναφέρω και ορισμένα παραδείγματα της δουλειάς που κάνουμε. Για να σχηματίσετε μια εικόνα. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας αναφέρω είναι ε, η δουλειά που κάναμε στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Υποστηρίξαμε την Προεδρία με τεχνικής φύσεως διαμεσολάβηση και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να φτάσουμε στην Ειρηνευτική Συμφωνία. Αυτό αποτελεί πολύ συγκεκριμένο πρακτικό τρόπο υποστήριξη μιας χώρας ε, σε μια κρίσιμη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τώρα τις γυναίκες δημοσιολαβητές επιτόπου, κάνουμε πολλή δουλειά στη Συρία, συνδέουμε το Συριακό Δίκτυο με το Δίκτυο στην Ιεμένη και συνεργαζόμαστε με το Βαρτσινρίφη και τον υποστηρίζουμε για να είμαστε σίγουροι ότι οι γυναίκες μπορούν να παίξουν πιο μεγάλο ρόλο στην εφαρμογή της συμφωνίας. Και ακόμη και σήμερα είχαμε μία συνάντηση με τη Φρεντερίκα Μογκερίνη και διαμεσολαβήτριες ε, από όλο τον κόσμο. Υπήρξε μία ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και ανταλλαγή εμπειριών για το τι σημαίνει να είσαι διαμεσολαβήτρια, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τις γυναίκες αυτές. Και ελπίζω ότι θα είδατε κάποια tweets ε, που ε, δημοσιεύτηκαν από αυτή την εκδήλωση σήμερα. Φυσικά, συχνά έχουμε συναντήσεις με τα κράτη-μέλη και καλούμε και το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις ε, με τους επαγγελματίες στον κλάδο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια κοινή προσέγγιση για την υποστήριξη της διαμεσολάβησης. Το αίτημα λοιπόν για τη διαμεσολάβηση και πρόληψη των σειράξεων αυξάνεται εκθετικά. Δυστυχώς θα έλεγα. Και επομένως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Σε Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό, αλλά και όχι μόνο, θέλουμε να είμαστε σε ηγετική θέση. Και πραγματικά βάζουμε τη δυνατά μας για να καταστεί εφικτό. Και να κλείσω μοιραζόμενος μία πρόκληση μαζί σας. Όπως ξέρετε, η διαμεσολάβηση και η πρόληψη των σειράξεων ε, πάντοτε γίνονται με έναν τρόπο πολύ διακριτικό και μερικές φορές είναι δύσκολο να δείξεις τις επιτυχίες σου και επιπρόσθετα υπάρχει και το θέμα της ανάθεσης. Δηλαδή, αν δεν συνέβη μια σύραξη, δεν έλαβε χώρα, πώς μπορείς να αποδείξεις ότι εσύ ήσουν αυτός που συνεισέφερε σε αυτή την επιτυχία, δηλαδή να μην ξεσπάσει αυτή η σύραξη. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα, δεν είναι μόνο δικό μας ε, πρόβλημα, αλλά είναι και πρόβλημα του Κοινοβουλίου αλλά και όταν συνομιλώ και με τον, ΟΣΑ, ΟΑΣΕ, συγγνώμη, με τα Ηνωμένα Έθνη, ε, όλοι ε, ασχολούνται με αυτό το θέμα ε, και θα πρέπει να ανταλλάξουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή τις εμπειρίες τους και μπορούν να πούνε, περνούν το σχάρι, εδώ έχω τέλεια παραδείγματα, δέκα τέλεια παραδείγματα, όπου μπορέσαμε να αποτρέψουμε μία σύραξη. Για να συνοψίσω, δεν τα έχω πάει και τόσο καλά με το χρόνο. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την έκθεση και για το σημαντικό σας έργο, για την πρόθεση της σημασίας της πρόληψης των σειράξεων και της διαμεσολάβησης. Και τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη για την πέμπτη επαιτειό του. Και να τονίσω πόσο σημαντική είναι για μας στο πλαίσιο της συνεργασίας τέτοια ιδρύματα όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη είναι απολύτως απαραίτητα αν ε, θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας και είναι απολύτως ε, βασική λοιπόν η συνεργασία μας με τέτοιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ όλους σας και τον τελευταίο μας ομιλητή. Καταρχάς, συνάδελφε, να πω ότι είμαστε, εορτάζουμε την πέμπτη επέτειο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη. Σήμερα το βράδυ στις 6.30 στον οίκο της Ευρωπαϊκής ε, Ιστορίας εδώ στο πάρκο Λεοπόλντ. Έχουμε ε, εκπροσώπους που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Ακούμε τον συνάδελφο. Ευχαριστώ Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλια. Όντως η Επιτροπή ΑΦΕΤ από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος προσπάθησε να παρουσιάσει όλο το πορτοφόλιο για, το, για την κλιματική διπλωματία. Έχουμε τα συμπεράσματα, συμβουλίου, το, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Έχουμε δύο για την κλιματική διπλωματία και ένα για την κλιματική διπλωματία και ένα για την διπλωματία του νερού. Και γι' αυτό μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε το τι έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει την έκθεσή μας και στον κύριο Κουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ε, την ολοκληρώσαμε πριν από λίγο καιρό και στη Χέλγα Σμιτ για την, ε, ε, για την δώσαμε την έκθεσή μας και στην Γερμανία. Εγώ μίλησα στην Γερμανία και θα μπει και στην ε, συνέλευση της διάσκεψης για την ασφάλεια στο Μόναχο την επόμενη φορά. Αυτό που κάναμε είναι να δείξουμε το τι γίνεται και από ποιες οπτικές το προσεγγίζουμε. Μιλήσαμε για την ε, γερμανική όθηση. Θα προσπαθήσουμε από κοινού με τη Σουηδία να πιέσουμε για να μπορέσουμε να ε, εμπλουτίσουμε το ΟΗΕ και να εντείνουμε την ε, γνώση και επιτόπου να βάλουμε και κάποιους μικρομηχανισμούς ώστε να μπορούμε ετησίως να ξέρουμε περισσότερα για το πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις εξελίξεις αυτό το ξεκίνησε η Σουηδία, τώρα αναλαμβάνει η Γερμανία ένα κομμάτι. Χέλκα Σμιτ μίλησε για το, για το δικό της κομμάτι και εγώ για την έκθεσή μας. Δύο ερωτήσεις έχω να θέσω. Ε, Γενικώ νομίζω ότι η κλιματική διπλωματία και η ε, δική μας η Επιτροπή έχει αφοσιωθεί σε αυτό, ελπίζω να το κάνει και η επόμενη θητεία, η επόμενη, το επόμενο κοινοβούλιο. Έχουμε αφοσιωθεί λοιπόν στο θέμα το ότι η κλιματική διπλωματία έχουμε, έχει, είναι ένα σημαντικό α, θέμα και έχουμε και τον οδικό χάρτη του Κατοβίτσε. Για να δούμε πώς μπορεί να, πώς μπορεί να και οι στόχοι του Παρισιού. Um, as you mentioned yourself, the climate is an important issue. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός γι' αυτό και αυτό έχει να κάνει και με το ερώτημα προς τον κύριο Φανής. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο μέσα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο να συμπληρώσουμε ε, το επίτευξη του στόχου για το 25%-30% για το κλίμα. Θέλουμε, είπατε κι εσεί, ε, δυνατότητε. Θέλουμε εμπειρογνώμονε. Τέσσερις άνθρωποι δουλεύουν στην ε, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων για το θέμα αυτό, για το κλίμα και την κλιματική διπλωματία. Θεωρείτε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα μονάδα, ας πούμε, μια νέα υπηρεσία συμπεριλαμβανομένη και αυτή που αναφέρατε, γιατί το κλίμα πραγματικά είναι πολύ σημαντικό παράγοντα για την κλιματική ε, διπλωματία. Όπω και ο μικρομηχανισμό που προσπαθούμε να, έχουμε στο, να εγκαταστήσουμε στον ΟΗΕ. Ίσως καλό θα ήταν να έχουμε κάτι αντίστοιχο και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη προσπαθούν να κάνουν κάτι, η Γερμανία, η Σουηδία α πούμε, αλλά επειδή η Γερμανία θα αναλάβει την Προεδρία, εσεί πώ πιστεύετε ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Thank you, And now... Ευχαριστώ εγώ. Ο Τσάρλ Στάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάπως διοικητικό είναι το θέμα μου. Ένας από τους υπαλλήλους εδώ μου είπε ότι ο υποψήφιος της CCR στο Συμβούλιο έφυγε από την Επιτροπή μάλλον λόγω διοικητικών προβλημάτων ε, εγώ δεν το ήξερα αυτό, είμαι και συντονιστή, αλλά δεν το γνωρίζω. Οπότε δεν ξέρω αν είχαμε τα τελευταία δυόμιση χρόνια ε, μέλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κρίμα. Δεν το γνώριζα. Θα, είχα, θα το είχα αναλάβει εγώ, αν το γνώριζα πιο πριν. Δεν ξέρω τώρα αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από τα οκτώ κρατημέλη που ασχολούνται με την ε, διαχείριση του ε, Ινστιτούτου. Από την προφορά σας, ε, κύριε Κίτινγκ, κατάλαβα ότι είσαστε από τη χώρα την οποία γνωρίζω πολύ καλά. Εμείς ακόμα εδώ είμαστε βέβαια, μάλλον θα πρέπει να έχουμε φύγει τρεις μέρες πριν. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Ίσως να μην είμαι καν εγώ εδώ. Μπορεί να είναι εδώ το ολόγραμμά μου. Όχι, όχι. Η Βρετανία προς το παρόν είναι ακόμα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μου λοιπόν το οποίο σχεδιάζεται και με την αυριανή συνεδρίαση με τον Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίο θα μιλήσει για τι μελλοντικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Εγώ είμαι από τους, ε, από τους Τόρι και είμαι ένας παλιός καλός ε, οπαδός του να παραμείνουμε στην Ένωση. Δύσκολος ο ρόλος μου. το θέμα της ε, διαμεσολάβηση ε, και της αντιμετώπιση των ε, συγκρούσεων δεν είναι από τα θέματα με τα οποία έχω ενεργώ ασχοληθεί, αλλά πραγματικά είναι εξαιρετική η δουλειά που έχετε κάνει για την Σομαλία, ας πούμε, μια χώρα που την ξέρετε πολύ καλά κύριε Κίτινγκ. Επίσης, τι γίνεται με την αντιμετώπιση τη πειρατεία. Αν το Brexit ε, αναστραφεί, έχουμε χάσει πάρα πολλές υπηρεσίες, πάρα πολλές αρχές, δυστυχώς. Αλλά η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, αν γίνει όντως το Brexit, βέβαια μπορεί να γίνει δεύτερο δημοψήφισμα, μπορεί να αναστραφεί, ακόμα είναι πολύ ρευστά τα πράγματα, και τώρα ακόμα ετοιμάζονται για ψηφοφορία στην Βουλή για να δούμε πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Το ΕΒ, λοιπόν πώς μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη δική σας την ε, υπηρεσία, με το δικό σας το Ινστιτούτο μετά τον Brexit, γιατί πραγματικά είναι ένας χώρος στον οποίο θα ήθελε να εμπλακεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα και όσοι θέλουν να αποχωρήσουμε το θέλουν αυτό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε πολύ καλή συνεργασία παρά την οδυνηρή αυτή και καταστροφική προοπτική και διαδικασία του Brexit. Thank you, Charles Claire Moody, please. Η Claire Moody. Ναι, ίσως χρειαζόμαστε μια ειρηνευτική διαδικασία και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά τέλος πάντων αυτό σχόλιο εν παρόδο. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Βανής για την επικοινωνιακή δουλειά που χρειάζεται να συνοδεύει πάντοτε τη δουλειά που σχετίζεται με την ειρηνευτική διαδικασία. Με μεγάλο ενδιαφέρον ε, παρακολούθησα και τον κύριο Κίτιν και τον κύριο Βανής, ιδίως όταν μιλήσατε για το πρακτικό έργο που επιτελείτε. Αναφερθήκατε και οι δύο λοιπόν στη σημασία που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία, στις ειρηνευτικές διαδικασίες και αναφερθήκατε συγκεκριμένα στη συνεργασία σας με ε, οργανώσεις γυναικών στην ε, Ιεμένη και στο Αφγανιστάν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, υπάρχουν τέλο πάντων πολλά παραδείγματα συμμετοχή των γυναικών στις συνευτικέ διαδικασίε. Και εγώ νομίζω ότι είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε. Γιατί πολλέ φορέ γίνεται λόγο για την ανάγκη να συμμετέχουν οι γυναίκε, αλλά Νομίζω ότι αυτό που έχει σημαντικό, αυτό που είναι σημαντικό είναι πώς πρακτικά τα παραδείγματα αυτά, οι περιπτώσεις όπου οι γυναίκες πραγματικά συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία, συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίτευξη της ειρήνης και χρειάζεται να το, να το διαφημίσουμε ότι πράγματι ήταν ένα στοιχείο για την υπέρβαση ή για την πρόληψη συγκρούσεων γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της βιωσιμότητας της όλης διαδικασίας η συμμετοχή των γυναικών σε αυτήν. Ευχαριστούμε. Άλλος ένας ε, συνάδελφος ε, από την Βρετανία, ο κύριος Κάβα. Ε, εργάζονται σκληρά σήμερα οι Βρετανοί. Ευχαριστώ, Ντέβιτ. Προφανώς εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί δεν θέλω επικάλυψη. Όμως πρέπει κανείς να γνωρίσει ότι κάθε προσπάθεια που κατευθύνεται προς την ειρήνη είναι θετική. Ο Τσάλς Τάνοκ αναφέρθηκε σε ένα θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ και εγώ. Ε, ακόμη και ως υπέρμαχος ε, του Brexit, εγώ ελπίζω να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν είναι σήμερα το θέμα μας. Ε, πρέπει να αναφερθώ. Άκουσα και από τον, τον Edward για το έργο που επιτελεί ο οίκος Ζαν Μονέ στην Ουκρανία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι αν πράγματι ε, θα δουλέψουμε προς την ειρήνη, ε, εγώ, ξέρετε, υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία απόψεων ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ΕΛΚ, σοσιαλιστές, ECR αν χρειάζεται να συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του οργανισμού, προφανώς και θα πρέπει όλοι να εκπροσωπούνται. Ε, ε, θα μπορούσε να υπάρχει και εκπρόσωπος από την ΚΟΕ. Βέβαια ξέρουμε ότι οι συνάδελφοι από την ΚΟΕ πιο πολύ ασχολούνται με, την, με τη Βενεζουέλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να τιμήσει τον τίτλο τη Ενωμένη στην Πολυμορφία, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσει ότι θα ακούγονται όλε οι φωνέ για κάθε ζήτημα. Και άκουσα βεβαίως τον Έλμαρ Μπρόκ που μίλησε ε, και χωρίς να διαφωνούμε, γιατί συμφωνούμε στον τομέα της Ουκρανίας, αλλά δεν γίνεται να μιλάει μόνο ένας ευρωβουλευτής όταν εκφράζεται η, η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ουκρανία. Χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία όσον αφορά την παρουσίαση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ακριβώ γιατί υπάρχει μια ε, πυκλομορφία και στι απόψει μας. Εγώ, για παράδειγμα, ε, έχω συγκεκριμένη άποψη για τη Σομαλιλάνδη ή θα μπορούσα να τοποθετηθώ σε συζητήσει και για τη Μογκαντήσου. Ε, ξέρετε ότι ε, θα μπορούσα ε, εγώ να λειτουργήσω ως κόκκινο πανί για εκπροσώπους της Σομαλίας. Ακριβώς γιατί είναι πολύ γνωστές οι απόψεις μου για την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει σε κάθε θέμα να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση, η δίκαιη, η θεμητή εκπροσώπηση όλων των απόψεων που εκφράζονται και εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακριβώς για να εξασφαλίζεται αυτό που λέει και το σύνθημά μας, ε, ενότητα στην πολυμορφία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμασούρ, που είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Κίτινγκ για το εξαιρετικό του έργο. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένος. Από ό,τι κατάλαβα, ξεκινήσατε λίγο πιο νωρίς τη συζήτηση. Δεν μπορούσα να ακούσω λοιπόν τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Θα έχουμε την δυνατότητα με την ευκαιρία ε, της, του εορτασμού της ε, πέμπτης επαιτίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ειρήνη θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε. Ο πρώτος ε, στόχος υλοποιήθηκε, ήταν η σύσταση ενός οργάνου ικανού να προβαίνει στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση κινητοποιώντας ε, προσωπικότητες, διαδικασίες, ε, όργανα και τεχνογνωσία για την ε, διατήρηση της ειρήνης ή για τη διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπόλεμων μερών και χρησιμοποιώντας τα καλύτερα της ευρωπαϊκής διπλωματίας με την ευρία του όρου κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συγκρίνουμε την ευρωπαϊκή διπλωματία με την αμερικανική, θα έλεγα, υπερβάλλοντα κάπω, ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, οι Αμερικανοί στέλνουν στρατό και κατόπιν διαπραγματεύονται, ενώ οι Ευρωπαίοι στέλνουν επιτόπου διπλωμάτε, γιατρού ε, ή και ανώκρανους. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη σε αυτό το πνεύμα έχει δημιουργηθεί έναν εξάρτητο όργανο από τα κράτη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αρκετά κοντά σε άμεση σύνδεση με την υπηρεσία εξωτερική δράσης για να μπορέσει να δώσει στα εμπόλεμα μέρη, αν φτάσουν σε συμφωνία από την αιγίδα του Ινστιτούτου, την εγγύηση να υπάρξει συνέχεια μια πολιτική υποστήριξη της Ένωσης. Ο δικός μας στόχος ήταν να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και όταν στέλνουμε διπλωμάτες, ΜΚΟ ή στρατιωτικούς επιτόπου ε, όχι ε, μόνο ε, να διαχειριστούν την κατάσταση, αλλά να διαβιβάζουν και την τεχνορωσία τους σε αυτούς που θα τους διδεχθούν και στην επόμενη γενιά. Γιατί αυτοί θα βοηθήσουν στο να αναδυθεί ένας, ένα κοινό πνεύμα, μια ευρωπαϊκή διπλωματία. Και πάλι με την ευρεία είναι του όρου, γιατί υπάρχουν κράτη που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Και το δεύτερο που θέλω να ξέρω είναι αν ο κύριος Κίτινγκ ε, έχει κατά νου κάποιες νέες εξελίξεις. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμασούρ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Για τον κύριο Κίτινγκ ήταν περισσότερες ερωτήσεις. Um, well, Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Στα σχολιά μου θα έπρεπε να πω ότι κάτι μοναδικό για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη είναι ότι είχε ένα συμβούλιο που αποτελείται από ευρωπαϊκά κράτη. Η κύρια σύμπραξή του, και δίκιο έχει ο Ρενέ, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είμαι πιο Ακριβή είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και συγκεκριμένα με την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Επίση συνεργάζεται στενά και με άλλα μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΔΕΦΚΟ, την Καμαδελτανίαρ και πολλού άλλου εταίρους. Αλλά η υπηρεσία εξωτερική δράση είναι ο κύριο εταίρο μα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τα κράτη-μέλη. Όμω, το θέμα είναι ότι πρόκειται για ένα εξάρτητο Ινστιτούτο, δηλαδή μιλάμε για μία μοναδική οντότητα. Η ιδέα είναι ότι να έχεις και τα πλεονεκτήματα ε, του Συμβουλίου που έχει διπλωματικό βεληνικές, διπλωματική επεύθυνση, αλλά να έχεις και την ε, ευελιξία την επιχειρησιακή ενό ανεξαρτήτου φορέα. Δηλαδή μπορείς να συνομιλήσεις με όλους, από τις κυβερνήσεις μέχρι με τους ανθρώπους που βρίσκονται επί τόπου και άμεσα ε, μπορεί να συμμετέχουν σε μία σύραξη και δεν προέρχονται περίπου χάρη από κυβέρνηση και μιλάμε και για μη παράγοντες. σε ό,τι αφορά την ερώτηση του Αρνελίτσα για την κλιματική διπλωματία. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Η δική μου παρατήρηση, και δεν έχω επεφελθεί και θα το κάνω μετά από αυτή την συνάντηση και θα εξετάσω τι κάνετε, αλλά η παρατήρησή μου στον τομέα αυτό και σε σχέση με το έργο μου στο Αφγανιστάν, στη Μέση Ανατολή, στη Σομαλία, στη Συρία είναι ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για το πώς υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή και ο για τους σπόρους. Δεν μιλάμε για γη, νερό, αέριο, πετρέλαιο. Καταλαβαίνουμε πώς όλα αυτά συνεισφέρουν ε, στη δημιουργία συγκρούσεων ε, και υπάρχει ένα αίσθημα δικίας επιτόπου. Αυτό που δεν κατανοούμε πλήρω ακόμα είναι πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, αυτή την ενόρεση για να προωθήσουμε το διάλογο και πιο θετικά αποτελέσματα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να εργαστούμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την κλιματική διπλωματία Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη, κάποιοι μιλούν για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια σε εύθραστα κράτη. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ε, τρόπος ε, για να συνενώσουμε τις ε, κοινότητες. Τώρα, τρίτον, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του Τσάρλ Στάνοκ για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Συμβούλιο του Ινστιτούτου έχει ρητά, με έχει ρητά εμφαρίνει να αναζητήσω περισσότερα μέλη για το Συμβούλιο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το Ηνωμένο Βασίλειο να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο αν το επιθυμεί. Αυτή είναι λοιπόν μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Έχω συναντηθεί με τον Ράλιστε Μπέρτε πριν δύο εβδομάδε και ήταν ιδιαίτερα πρόθυμο και έδωσε την εντολή στους υφισταμένους να εξετάσουν ε, την ε, δυνατότητα αυτή. Βέβαια έχει αναχωρήσει από τη θέση αυτή και όπως έλεγα η Ελβετία είναι στο Συμβούλιο, δεν ξέρω αν ε, το είπα ή όχι ήθελα να το πω και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι κάποιες χώρες δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν στο μέλλον να είναι, αλλά έχουν πολλά να προσφέρουν στον τομέα αυτό. Και πράγματι, όταν πήγα στο Βερολίνο και στο Παρίσι, στη Στοκόλμη, στη Βαρσοβία και αλλού, υπάρχει ουσιαστικά ένα αίσθημα ε, λύπης ότι μπορεί στο μέλλον να μην έχουμε τόσο διαθέσιμη την τεχνογνωσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Στούτο για την Ειρήνη μπορεί να είναι από τους τρόπους ε, να το δισταθμίσουμε την απώλεια αυτή. Για τις ερωτήσεις ε, του κυρίου Λαμασούρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτα δίκιο ότι η γνώση που κερδίζεται από την πρόληψη και την επίλυση των σειράξεων θα πρέπει ουσιαστικά ε, να χρησιμοποιηθεί και να αντελαχθεί. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο στον τομέα αυτό όπως θα κάνουμε τώρα. Αλλά δεν είναι σημαντικό να τα κάνουμε μόνο εμείς, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά και μέσα από όλα όργανα. Κάτι που παρατήρησα είναι ότι σε ορισμένες ε, χώρες κεντρικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το θέμα της πρόληψης των συγκρούσεων επιβιώνει των εκλογών ενώ σε άλλες ε, χώρες ξανεμίζεται και εξαρτάται το χάρη από τη σύσταση των επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων, το προσωπικό που τις ε, στελεχώνει από τους ακαδημαϊκούς κτλ. Όμως θα θέλαμε να εξετάσουμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε ότι η διαχείριση της γνώσης δεν εξανεμίζεται. Και κάτι που δεν ανέφερα, για να κλείσω, είναι το εξή. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο υψηλών αξιωματούχων που παρέχουν συμβολές ε, παγκοσμίω. Δεν είναι όλοι Ευρωπαίοι και είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να επωφεληθούμε από μια τεράστια πρακτική εμπειρία ανθρώπων οι οποίοι έχουν συμμετέχει σε ελληνές διαδικασίες και σε διαδικασίες διαλόγου, έχουν ε, αναλάβει διαδικασίες διαμεσολάβησης και έχετε δίκιο. Πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο το πώς θα ανταλλαχθεί αυτή η εμπειρία μεταξύ αυτών, αλλά και πώς όλοι μπορούν να επωφεληθούν και μεταξύ κυβερνήσεων μερικές φορές ε, είμαστε κολλισμένοι σε ένα πρόβλημα μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά αν θες να επιλύσει συγκρούσει, πρέπει να συμμετέχουν και άλλοι φορεί. και βουλευτέ, παραδείγματο χάρη, και επιχειρηματικοί παράγοντε, ε, ομάδε, θρησκευτικέ, πολλοί άνθρωποι και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ότι οκτώ κυβερνήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν ε, Κρηματοοικονομική βοήθεια Βέλγιο, Φιλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ελβετία, Σουηδία. Ναι, και έχουμε τρεις ακόμη που ενδιαφέρονται στο να συμμετέχουν. Και κάτι που πρέπει να πω ακόμη είναι ότι κάποιες κυβερνήσεις που δεν είναι στο Συμβούλιο και μας δίνουν χρηματοδότηση για συγκεκριμένες δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη Ερβηγία κάτω χώρες. Έχουμε λάβει υποστήριξη από αρκετέ χώρες που για διάφορους λόγους δεν θέλουν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο, αλλά τους αρέσει η δουλειά που κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία ερωτήματα. Η πρώτη ερώτηση για την κλιματική διπλωματία του κυρίου Λίτς. Ναι, έχετε απολύτως δίκιο. Υπάρχει όντως ε, αύξηση της προσοχής που δίνουμε στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική διπλωματία, ο Μάικολ σωστά είπε ότι πρέπει να κατανοήσουμε πώς να προσεγγίσουμε ωστόσο το θέμα αυτό. Η κλιματική διπλωματία είναι το ίδιο με το να δούμε ας πούμε τον ανταγωνισμό για τη γη, ξέρουμε, στην, είναι βασική, ε, βασικός λόγος σύραξης στην Αφρική ας πούμε, είναι κάτι τελείω άλλο. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και εγώ θα με ενδιαφέρε πραγματικά να δω το έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται. Και βεβαίως γι' αυτό πρέπει να έχουμε και περισσότερο προσωπικό. Χρησιμοποιούμε ε, πολλούς δείκτες για το σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης ε, για να μπορούμε να προβλέψουμε πού υπάρχει ή πού θα υπάρξει μια βίαιη σύραξη στο μέλλον. Και αυτό πραγματικά είναι καινοτόμος προσέγγιση. Έχετε δίκιο, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Κάνουμε πιο πολλά από ό,τι κάναμε πριν από χρόνια. Ε, είπατε ότι είναι τέσσερι άνθρωποι που δουλεύουμε. Πριν από κάποια χρόνια δεν είχαμε κανέναν. Ε, οπότε είναι και αυτό μια βελτίωση. Ελπίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει και θα μπορέσουμε βεβαίω πάντα να είμαστε σε επαφή και σε ανταλλαγή απόψεων μαζί σα. Το θέμα είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο ότι ήταν ε, πραγματικά ε, παράδειγμα, υπόδειγμα με την αντίστοιχη υπηρεσία του για την αντιμετώπιση των ε, σειράξεων. Το να βλέπουμε τώρα το, το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι σε τροχιά αποχώρησης είναι πραγματικά λυπηρό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ε, την, άποψη, την συνεργασία που έχουμε με την υπηρεσία τυποποίηση, γιατί πραγματικά έχουν ατελείωτη τεχνογνωσία και εμπειρία. Προσπαθούμε λοιπόν και εμεί στη φάση αυτή να δούμε ακόμα και μετά τον Brexit πώ θα μπορέσουμε να, δούμε, να έχουμε καλύτερε εργασιακέ σχέσει. Η κυρία Μούντι μίλησε για την επικοινωνία. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να κάνω να πω οτιδήποτε. Καμιά φορά είμαστε, ξέρετε, λίγο συντηρητικοί, λέμε ότι είναι λίγο διακριτική η δουλειά που κάνουμε, αλλά μπορούμε σίγουρα να κάνουμε περισσότερα. Αυτό σίγουρα θα το έχουμε υπόψη μας. Αυτό επίσης που μπορώ να ε, μοιραστώ μαζί σας είναι ότι στην έκθεση που ε, μάλλον στα πλαίσια τη ε, μεταρρύθμιση που κάνουμε, είναι ότι έχουμε μια νέα υπηρεσία που θα ασχολείται με τα διδάγματα και με την τεχνογνωσία. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία θα μελετά το τι έχουμε επιτύχει, τι μπορούμε να μάθουμε από όσα έχουμε κάνει και πώς μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε λίγο περισσότερα, πώς μπορούμε να τα γνωστοποιήσουμε καλύτερα στον κόσμο, στα, πράκτη, στα κράτη-μέλη, στους ανθρώπους που δουλεύουν επαγγελματικά, πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στο διάλογο που κάνουμε με τον ΟΗΕ, με τον ΩΣΑ, με την Αφρικανική Ένωση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες. Η επικοινωνία λοιπόν και η διαχείριση της γνώσης θα είναι πραγματικά ψηλά στην ατζέντα μας για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Edward, πραγματικά ήταν πολύ καλή η συζήτηση αυτή. Και δείχνει ότι έχουμε πολλές ε, δυνατότητες ε, για να πετύχουμε σε πολλούς τομείς πολύ καλά αποτελέσματα. Διαμεσολάβηση, αντιμετώπιση συγκρούσεων κτλ. κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί μπορούμε να μάθουμε ημένα από τους δε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε ο συνάδελφός σας για την συνεργασία των πολιτικών ε, ομάδων του Κοινοβουλίου και να πάρουν μέρος στις διάφορες ε, προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η ιδέα αυτή καλή είναι γενικώ. Αλλά ειδικώ να πω ότι η εργαζο... οι ομάδες εργασίας της ΑΦΕΤ είναι το σημείο που μπορούν η κάθε πολιτική ομάδα να, μπορεί η κάθε πολιτική ομάδα να εκφράσει την άποψή τη. Όλα συζητούνται εκεί, είναι συμπεριληπτική η διαδικασία. Αλλά μετά πάμε στην διαμεσολάβηση αυτή καθ' αυτή. Και εκεί πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί στην προσέγγιση μα. Πρέπει να επιλέξουμε αυτούς που θα κάτσουν γύρω από το τραπέζι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες σε αυτό το τραπέζι. Πρέπει να σκεφτούμε πρακτικά εκείνη τη στιγμή. Και οι ε, ομάδες αυτές της διαμεσολάβησης ούτως ή άλλως, ούτως ή ε, αναφέρονται πίσω στην ε, ε, ομάδα της οποίας ηγείται ο κύριος Μακάλιστερ και η Λίντα Μακάνον. Και μπορούν να ακουστούν και εκεί οι απόψεις και τα αποτελέσματα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δουλειά και στο μέλλον. Τώρα για τη Βόρειο Μακεδονία ε, εκπροσωπείται το ΕΛΚ, εκπροσωπείται το ΑΛΔΕ και, το, ε, και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις ο εισηγητής θα πρέπει να, να παρίσταται στις διαπραγματεύσει. Και αν υπάρχει τώρα κάποιος που έχει κάποια ειδικότητα, κάποια συγκεκριμένη γνώση, εξειδικευμένη, και αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη όταν ξεκινά να συστήνεται αυτή η διαπραγματευτική ομάδα. Η ιδέα λοιπόν γενικώ είναι καλή, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές, λίγο πιο πρακτικοί στην προσέγγιση μας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Άλλος κανείς, άλλα σχόλια, παρατηρήσεις. Από εδώ κάποιος να θέλει να προσθέσει κάτι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους και τους τρεις προσκεκλημένους. Ελπίζω να γιορτάσετε ευχάριστα. Μέσα σε μισή ώρα θα ξεκινήσουν και οι εορτασμοί. Αυτά για σήμερα από μας. Κλείνουμε τη συνεδρίαση και θα τα πούμε αύριο στις 9 με τους ε, προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Καλό απόγευμα σε όλους.